Welcome everybody. Καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσει η συνεδρίασή μας και θα μιλήσω σουηδικά. Hej och välkomna till eh, det här. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Μόλις είχαμε συνεδρίαση των συντονιστών. Επομένως ολοκληρώσαμε το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης και πάμε στα άλλα. Σημείο 2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να σας αναφέρω μια αλλαγή. Το σημείο 7 η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεταφερθεί. Δεν μπορούμε να το εξετάσουμε σήμερα, θα πρέπει να το εξετάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Με αυτή την αλλαγή λοιπόν νομίζω ότι εγκρίνεται η μερίσχια διάταξη. Προχωράμε στο σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 27ης Μαρτίου του 2012. Προτείνουμε την έγκρισή τους. Προτείνουμε και την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 17ης και της 18ης Δεκεμβρίου του 2012. Επόμενο σημείο της ημερικής διάταξης είναι το σημείο 5, οι ανακοινώσεις του Προέδρου. Το μόνο που θα ήθελα να σας ανακοινώσω σήμερα είναι ότι έχουμε διερμηνία από 12 γλώσσες και προς 12 γλώσσες. Δεν είναι όλες οι γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι πολλές. Και θέλω να καλωσορίσω και την ομάδα των επισκεπτών. Στο βάθος της αίθουσας. Είναι προσκεκλημένη του μέλους της κυρίας Σιλβί Γκυγιόν, φοιτητέ του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών της Γαλλίας. Καλώς ορίσατε. Σας καλωσορίζουμε θερμά. Στη συνέχεια, ως προς το σημείο 5, θα ήθελα να κάνω μια τελευταία παρατήρηση. Ενδεχομένως γνωρίζετε ότι υπάρχει ένας κανόνας στο θεσμικό μας όργανο το οποίο ορίζει ότι δεν μπορεί το προσωπικό να δουλεύει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα για περισσότερα από ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών και θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν εσωτερική κινητικότητα. Έχουμε λοιπόν ένα, ε, κάποιον που έχει φτάσει σε αυτή την προθεσμία, τον κύριο Σόλταν Πέτο, ο οποίος ε, εργάζεται εδώ με μας εδώ και αρκετό καιρό και θα πρέπει να αλλάξει τμήμα. Λυπούμε πολύ που πρέπει να φύγετε. Έχετε κάνει πολλά για την Επιτροπή μας. Μας έχετε παρουσιάσει τη δουλειά σας με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό. Είστε πάντοτε χαρούμενος. Ε, δείξατε ότι θεωρείτε ότι πάντοτε όλα είναι δυνατά και όλα μπορούν να γίνουν. Δουλέψατε πάρα πολύ σκληρά. Νομίζω ότι σας εκτιμούν βαθύτατα όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Εγώ προσωπικώς εκτιμώ ιδιαίτερο στη δουλειά σας. Συνεργάστηκα μαζί σας σε πολλούς τομείς κατά τη σύνταξη των δικών μου εκθέσεων, στις οποίες εσείς συμβάλλατε τα μάλα και με βοηθήσατε όχι μόνο εμένα αλλά και άλλους ε, σε πολλές και διαφορετικές περιστάσεις. Είστε χαρούμενος, έχετε χιούμορ, είστε επαγγελματίε, είστε ε, ικανός και σας αρέσουν και οι Depeche Mode, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα. Νομίζω ότι είναι φυσικός. Όποιον αρέσουν οι Depeche Mode είναι σίγουρα καλός και στη δουλειά του. Νομίζω ότι είστε ένας πολύ πολύτιμος ανθρώπινος ε, πόρος, εκτός του ότι είστε και φαν των Depeche Mode. Κρίμα που σας χάνουμε. Αλλά παραμένετε βέβαια στο ίδιο θεσμικό όργανο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε άλλο τμήμα. Ίσως να έχουμε την ευκαιρία πάλι να μοιραστούμε τα των Depeche Mode άλλη φορά ή σε κάποια άλλη περίσταση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν ήξερα αν έπρεπε να το αναφέρω και να το μαρτυρήσω στους άλλους πόσο πολύ αγαπάτε τους Depeche Mode. Ήθελα τους τίτλους πολλών τραγουδιών των Depeche Mode να βάλω στην αποχαιρετιστήριά μου αυτή η ομιλία προς εσάς σήμερα, αλλά δεν τα κατάφερα. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και καλή συνέχεια στο έργο σας. Πάμε τώρα στο σημείο 6 Ανακοινώσεις του Προέδρου για άλλο θέμα όμως, για τις συστάσεις των συντονιστών της 21ης Ιανουαρίου του 2013. Δεν έχουν υπάρξει αιτήματα για αλλαγές σε αυτές τις συστάσεις, επομένως εγκρίνονται οι συστάσεις αυτές. Το 7 θα το εξετάσουμε κάποια άλλη στιγμή και γι' αυτό πάμε τώρα στο 8. Κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στην ε, συντάκτρια της νομοδότησης, Μότσα, Κλέβα και Κούτς από τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ, ήσασταν ακριβώς μπροστά μου και δεν σας είδα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όντως και εμένα μου αρέσουν πολύ οι Depeche Mode. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό το θέμα. Ας προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε. Συντέταξα μια γνωμοδότηση για την κοινωνική στέγαση στην ΕΕ. Βασική ε, συντάκτρια γνωμοδότηση είναι η Επιτροπή Θεμάτων Απασχόλησης, επί τη ουσία, δηλαδή. Ποτέ δεν υπάρχει χώρος σε μία γνωμοδότηση να συμπεριλάβει κανείς όλα όσα θα ήθελε. Ας τη θεωρήσετε τη γνωμοδότησή μου ως μία ραχοκοκαλιά και το ψαχνό σε αυτή τη ραχοκοκαλιά θα το γεμίσουν οι συνάδελφοι στην Επιτροπή για την απασχόληση και με βοήθησαν σε όλη αυτή τη δουλειά και οι σκιώδεις εισηγητές που συνεργάστηκαν μαζί μου όλο και πολύ περισσότερες είναι οι γυναίκες που διαβιούν σε κατάσταση φτώχειας από ότι οι άνδρες και λόγω των μισθολογικών ανισοτήτων και λόγω των διαφορών των φύλων και του χάσματος που υπάρχει μεταξύ αυτό. Και αυτό είναι πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2010 το 24% περίπου του συνόλου των γυναικών βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας, εξού και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό οφείλεται και στην κρίση την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και στις εξελίξεις της Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, το, οι οποίες είναι και οι συνέπειες, αν θέλετε, της κρίσης. Η κρίση είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερο ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες. Λόγω του χαμηλού εισοδήματος είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος για τις γυναίκες να διαβιούν σε μη ασφαλή και μη υγιή περιβάλλοντα. Θέλω να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας ε, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τις μόνες μητέρες, για παράδειγμα, Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι έχουμε 7 φορές περισσότερες μόνες μητέρες από μόνους πατέρες. Αυτές είναι, αυτά είναι στοιχεία τα οποία διάβασα πολύ προσφάτως. Εξού και θα πρέπει πιστεύω να τους δοθεί προτεραιότητα κατά την παροχή κοινωνικής κατοικίας. Έχω συμπεριλάβει όμως και άλλες ε, κοινωνικώς ευπαθείς ομάδες στη δομοδότησή μου, τους μετανάστες, τις, ε, τις μετανάστριες, τα άτομα με αναπηρία, γυναίκες από μειονοτικές ομάδες και ηλικιωμένοι. Νομίζω ότι είναι καλό να είναι κάπως καλύτερα και περισσότερο εστιασμένη η γνωμοδότηση αυτή. Καλούμε τα κράτη-μέλη να στηρίζουν τις γυναίκες για την επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας και παρέχοντας τις απαραίτητες συνθήκες για την συμφιλίωση οικογενειακής, προσωπικής και επαγγελματικής ε, ζωής. Αυτό είναι πάντοτε θέμα που απασχολεί τη δική μας Επιτροπή. Και τέλος, ε, θέλησα να δώσω περισσότερη σημασία στα θύματα της οικιακής βίας, τα οποία μένουν σε αυτό το νοσηρό περιβάλλον, κυρίως λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων. Και θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβασή τους σε μια κοινωνική κατοικία, η οποία θα είναι προσιτή οικονομικά. Θέλω, θα ήθελα να υπάρξει ξεχωριστή παράγραφος για αυτό. Και τέλος, ε, καλούμε τα κράτη-μέλη να διενεργούν αναλύσεις με βάση το φύλλο, ως μέρος όλων των ε, πολιτικών και ότι τα δεδομένα πρέπει να αναλύονται κατά φύλλο και πρέπει να υπάρξει περισσότερη έρευνα. Τα κράτη-μέλη αντιλαμβάνονται το όρο, τον όρο κοινωνική στέγαση με τελείως διαφορετικό τρόπο το καθένα. Δεν ήθελα να μπω σε αυτό το θέμα. Συμμετείχα στη συζήτηση τη σχετική που έγινε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιλήφθηκα ότι πραγματικά κάθε κράτο μέλο ερμηνεύει διαφορετικά τον όρο κοινωνική στέγαση. Δεν θέλησα να μπω λοιπόν, σε αυτή την τεράστια συζήτηση. Προτίμησα να επικεντρώσω τον ενδιαφέρον μου στι γυναίκε και στη γνωμοδότησή του, γιατί αυτό μα αφορά άλλωστε. Αλλά αδειμονώ για περαιτέρω συνεργασία με του κοιόδη συζητητέ και του υπολείπου συναδέλφου και συναδέλφου γυναίκε της Επιτροπής μας κατά τους επόμενους μήνες, ούτως ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα λόγος στους συναδέλφους. Στους συναδέλφους. Uh, thank you, Chair. I thank Rapporteur. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά της και συμφωνώ με τις περισσότερες από τις απόψεις που εκφράζει στη γνωμοδότηση. Δεδομένου ότι στην Ευρώπη έχουμε 7 φορές περισσότερες μητέρες μόνες από ότι πατέρες και επειδή οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση θα πρέπει να τους να τις προστατεύσουμε περισσότερο. Θα πρέπει να τους δοθεί προτεραιότητα για μια κοινωνική, κοινωνικού τύπου στέγαση η οποία να μην είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους στέγαση αυτή τη στιγμή και σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Σε πολλά κράτη-μέλη προβλέπεται κοινωνική στέγαση, αλλά με τιμές ιδιαίτερα υψηλές. Το επίπεδο των τιμών είναι παρόμοιο με το τι συμβαίνει στην αγορά ακινήτων γενικότερα. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστεί πρόσβαση στην ε, αξιοπρεπή ε, στέγαση και κατοικία. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Undrar om det är så att någon från kommissionen skulle vilja ta ordet? Ε, υπάρχει κάποιο άλλο που θα ήθελε να παρέμβει. Παρακαλώ. Καλησπέρα σα. Λέγομαι Γιώργο Ζόμπερέκερ από την Γενική Διεύθυνση Εργασία. αλλά ενώ υπάρχουν περισσότερε ε, μόνε μητέρε από ότι πατέρε, 7 φορέ περισσότεροι, είναι περισσότεροι άστεγοι άντρε από ότι γυναίκε. Θα πρέπει λοιπόν ε, στο πλαίσιο τη κοινωνική στέγαση να σκεφτούμε μια λύση και για αυτή την πτυχή. Somebody else? Κάποιος Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, ο λόγος και πάλι στην εισηγητρία. Ευχαριστώ. Αναφέρθηκα στις μόνες μητέρες, τις άγαμες μητέρες, γιατί σε κάποια μελέτη το εντόπισα και θεώρησα ότι είναι σημαντικό. Καλωσορίζω πάντως όλα τα σχόλια και νομίζω ότι όποια συνεισφορά θα εμπλουτίσει την σημερινή γνωμοδότηση. Αν υπομονώ λοιπόν για τη συνεργασία σας τις ερχόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Uh, verkar inte vara som att eh, det finns någon mer som vill sätta upp sig. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Οπότε, να σας ανακοινώσω τις προθεσμίες. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, 25 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα. Ενώ η γνωμοδότηση θα ψηφιστεί στην Επιτροπή μας στις 20 Μαρτίου. Η Επιτροπή Απασχόλησης θα ψηφίσει στις 23 Απριλίου. Μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε το σημείο αυτό και να περάσουμε στο επόμενο. Το 9. Αναπτυξιακή στόχη της χιλιετίας. Ορισμός του πλαισίου μετά το 2015. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ντελβό, την εισηγήτρια. I don't see Mrs. Delvaux, but... Uh, Δεν βλέπω την κυρία Ντελβό. Υπάρχει κάποιος άλλος από το ΕΛΚ που θα ήθελε ξανά με το στις να πάρει το λόγο. Κυρία Μπάουερ. Βλέπω ότι ανυπομονείτε και κάνετε νεύματα. Κάποιος κλώδης εισηγητής, εισηγήτρια, θα ήθελε το λόγο. Ναι, κάποιος άλλος βουλευτής. Οποιοςδήποτε, κάποιος. This is really strange. Πραγματικά παράξενο. Προφανώ όλοι είναι ικανοποιημένοι με την έκθεση. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Δίκιο έχετε. Normally everything takes much longer than... Κάποιος από την Επιτροπή θα ήθελε το λόγο. Σας παρακαλούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή είναι πάντοτε ετοιμόλογη και επιθυμεί να παρέμβει. Γι' αυτό να κάνω κι εγώ ένα-δυο σχόλια για το σχέδιο νομοδότησης που είχα την ευκαιρία να το διαβάσω. Καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον σα για το τι θα γίνει με του αναπτυξιακού στόχου μετά το 2015 και ο Επίτροπο Πίμπαλξ ήρθε δύο φορέ στην Επιτροπή Ανάπτυξη για να συζητήσει μαζί του τα θέματα αυτά και να αναπτυχθεί ο σχετικό διάλογο. Καλωσορίζουμε το σχέδιο γνωμοδότηση. Υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία βρίσκουμε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα, κυρίω το ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη εξουσία στι γυναίκε ω ένα μοχλό για την πρόθεση τη ανάπτυξη και ότι χρειάζεται και ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση για την ε, τόνωση των στόχων. Νομίζω ότι αυτές ήταν χρήσιμες συνεισφορές. Η ισότητα των φύλων είναι μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απασχολεί την ε, συζήτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ένα αυτόνομο θέμα, αλλά και ως ένας ε, τρόπος για να ενισχυθεί η ανάπτυξη για μετά το 2015. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια προετοιμασία μια ανακοίνωση για το τι θα γίνει μετά το 2015 με το σχετικό πλαίσιο και του αναπτυξιακού στόχου. Και σε αυτό το επίπεδο πιστεύουμε ότι η κρίση τη φτώχεια θα πρέπει να παραμείνει μια από τι βασικότερε προτεραιότητε τη μελλοντική μα ατζέντα. Ότι θα πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω του στόχου τη χιλιετία που ήδη υπάρχουν, αλλά και να ενισχύσουμε σημεία τα οποία ήταν αδύναμα ή έλειπαν από το σημερινό πλαίσιο. Όμως δεν θα πρέπει να βιαστούμε αυτή τη στιγμή ε, σε αυτή τη χρονική φάση να κάνουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωση, γιατί οι συζητήσεις είναι ακόμη πρώιμες. Στον ΟΗΕ οι σχετικές συζητήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί και νομίζουμε ότι το κατά πόσον θα επιτύχει ο καθορισμός των στόχων μας και η μελλοντική μας ατζέντα είναι το κατά πόσον θα αναλάβουν και την ευθύνη οι χώρε που περισσότερο ε, πρέπει να δράσουν εδώ. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά και ο ΙΕ, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξουν τις χώρες αυτές τις προσπάθειές τους. Δεν θα πρέπει όμως τώρα να είμαστε πολύ δεσμευτικοί στην αρχή της διαδικασίας. Η ανακοίνωση πρόκειται να εγκριθεί στα τέλη Φεβρουαρίου και ελπίζουμε του ερχόμενου μήνες να έχουμε και άλλε συζητήσει με το Κοινοβούλιο του θέματο αυτού. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο μόνος και ο δισεισηγητής που παρευρίσκεται είμαι εγώ ίδιο. Θα σχολιάσω λοιπόν κι εγώ, γιατί οι στόχοι της χιλιετίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για πολλούς διαφορετικούς τομείς. Η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι κέρια για το μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να συμβάλλει το Κοινοβούλιο μας σε αυτήν την διαδικασία. Ελπίζω ότι οι μελλοντικοί στόχοι της χιλιετίας θα περιλαμβάνουν τη διάσταση ισότητας ανδρών και γυναικών. διαπιστώνουμε ότι συνήθως οι γυναίκες πλήττονται από τη φτώχεια ή την επισφάλεια, την εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και αυτή η διάσταση της ισότητας των φύλων στους στόχους της χιλιετίας, αλλά θα πρέπει και οι υπόλοιποι στόχοι να συμπεριλαμβάνουν αυτή τη διάσταση. Όταν μιλάμε λόγω χάρη για την εκπαίδευση και την παιδεία, είναι καθοριστική σημασία να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια να εκπαιδεύονται. Ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει συνολικά την κοινωνία. Πρέπει λοιπόν η ισότητα ανδρών και γυναικών να είναι ένα θέμα που να αφορά όλους τους τομείς, οριζόντιο. Βεβαίω είναι και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν δεν πετύχουμε την ισότητα μεταξύ των φύλων, δεν πρόκειται να υπάρξει πραγματικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πώ θα τοποθετηθούν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνεί οργανισμοί όπω ο ΟΗΕ είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και η δική μα Επιτροπή αλλά και η Επιτροπή για την Ανάπτυξη θα πρέπει να εργαστούν για να προωθήσουν τα δικαιώματα των γυναικών. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μπάουερ τώρα. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά, θα ήθελα να στήσω συγγνώμη, γιατί πιο πριν μιλούσαμε για την ε, ψηφοφορία, την αυριανή, και έχασα λίγο την προσοχή μου, αφαιρέθηκα. Να τονίσω τη σημασία που έχει το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε σε αυτό το στάδιο των εργασιών μα ε, όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες, διότι ως μέλος της αντιπροσωπείας ΑΚΕ, πολλές φορές παρατηρώ ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρά, απίστευτα προβλήματα. Βρισκόμαστε σε... Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τα ζητήματα των γυναικών. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί κατά πολύ η θνησιμότητα των ε, γυναικών που γεννάνε στην υποσαχάρια Αφρική. Τα νούμερα ωστόσο παραμένουν υψηλά. 350.000 γυναίκες κάθε χρόνο είναι θύματα της ελάθος υγειονομικής περίθαλψης και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να προωθήσουμε και να στηρίξουμε την εκπαίδευση των μεών. Πιστεύω πως πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. κατά τη διάρκεια του επόμενου προγράμματος μας και έπειτα μία πάρα πολύ άσχημη κατάσταση σε ορισμένες χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής είναι και η βία ενάντια στις γυναίκες. Και εκεί παρατηρούμε πως υπάρχουν πάρα πολλοί υψηλοί αριθμοί γυναικών θύματων οικογενειακής βίας, σεξουαλικής βίας. Πολλές χιλιάδες. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας και θα έπρεπε να ασχοληθούμε με αυτό. Τώρα, εξεπλάγει από το εξή. Σε μία χώρα που δεν θα ήθελα να κατονομάσω, υπάρχει ένας αγώνας καταπολέμησης της διαφθοράς. Αλλά παρά τις προσπάθειές μας, η διαφθορά δεν θα εξαλειφθεί πλήρως. Αυτό που θα βοηθούσε είναι να ασχοληθούμε με τον τομέα της υγείας, με τον τομέα της ευβίας των γυναικών. Διότι πραγματικά είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση εκεί στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω είναι ότι θα μπορούσαμε να ξαναδούμε τις προτεραιότητές μας στην αναπτυξιακή πολιτική από την σκοπιά της ισότητας των φύλων. Ευχαριστώ. Yes, thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η κυρία έχει το λόγο. Ε, ζητώ συγγνώμη που έφτασα αργά κατά τη διάρκεια της επαρέμβασης της κυρίας Μπάουερ. Θα είμαι σύντομη. Κοίταξα το σχέδιο γνωμοδότησης και νομίζω πως όλα είναι εντάξει. Όμως θα ήθελα αυτή η Επιτροπή να πάει λίγο πιο πέρα και να είναι λιγότερο διστακτική, διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια μιλούμε και καταδικάζουμε αυτά που μόλις περιέγραψε η κυρία Μπάουερ. Και πιστεύω πως έχουμε μείνει πολύ πίσω όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα, την υγεία και τη σεξουαλική βία. Έχει... Δεν υπάρχει πολιτική θέληση, πιστεύω. Και να τονίσω ότι εμείς λειτουργούμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά, διότι εάν κάποιο άλλο κομμάτι του πληθυσμού δεν απολάμβανε πλήρως ή του στερούνταν τα, τα βασικά του δικαιώματα. Εμεί θα κάναμε εισβολή στη χώρα, στρατιωτική επέμβαση. Αλλά τώρα αυτό δεν ισχύει. Λέμε εντάξει, ωραία, τι άσχημα που υποφέρουν οι γυναίκε, είναι λυπηρό, κρίμα. Και να σα δώσω και ένα παράδειγμα. Στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μία ρήτρα, το No Abortion Clause, ρήτρα μη αμβλώσεων. όπου όχι μόνο δεν παρέχονται κονδύλια και δεν παρέχεται βοήθεια για γυναίκες ε, για, που, έχουν, ε, που έχουν βιαστεί και έχουν μείνει μετά έγκυες να κάνουν αμβλώσεις, αλλά υπάρχει εντολή να αποσιωπήσουν το ζήτημα. Πολλές φορές, πολλές γυναίκες, ε, στο Κονγκό για παράδειγμα, πέφτουν θύματα βιασμού και, εμείς, και αρνούνται μετά τα νοσοκομεία να τους παρέχουν υπηρεσίες άμβλωσης και εμείς σιωπούμε. Δεν είναι αρκετό να ψηφίζουμε το ένα ψήφισμα μετά το άλλο. Πρέπει να στηρίξουμε πολιτικές που θα υποστηρίζουν τις γυναίκες και θα βοηθούν τις γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα χαιρέτιζα ένα ψήφισμα το οποίο θα ενδυνάμωνε τα δικαιώματα των γυναικών και θα είχε πράξεις και όχι μόνο λόγια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ιντφέλτ. Αρχίσαμε με μια παρέμβαση της Κομισιόν, ζητήσαμε από την Επιτροπή να πει κάτι. Στην αρχή είχαμε πάρα πολύ ησυχία και τώρα άρχισαν να έρχονται όλοι. Τώρα ήρθε και η συγγήτρια. θα μιλήσει στο τέλος, κανονικά θα έπρεπε να είχε μιλήσει στην αρχή, αλλά δεν πειράζει, ακούσαμε όλους τους συναδέλφους και τώρα έχει η το λόγο. κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Πολλές επιτροπές αρχίζουν την ίδια ώρα. Είχα ήδη εξηγήσει το στόχο αυτής της έκθεσης το πρόγραμμα των στόχων για την χιλιετία που ξεκίνησε το 2000 θα ολοκληρωθεί περίπου το 2015. Επομένως, αυτή τη στιγμή ε, εξετάζονται εκ νέου οι ορισμοί για τους, στόχους, τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή για την Ανάπτυξη και θα πρέπει να λάβει υπόψη τις δικές μας συστάσεις για την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών και ούτω καθεξής. Δύο αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας στρέφονται γύρω από τις γυναίκες, στόχος 3 ε, προώθηση ισότητας φύλων κλπ. και στόχος 5 βελτίωση της υγείας των ε, μητέρων. Και παρά τις ε, προόδους που έχουν γίνει, εκατέρωθεν μένει πολλή απόσταση που θα πρέπει να διανυθεί για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η πρόοδος λοιπόν φαίνεται σε αυτό το πίνακα που έχει σκιαγραφηθεί και αυτός ο πίνακας παρουσιάζει πάρα πολύ λες ελλείψεις, π.χ. στο ποσοστό των κορισιών που πηγαίνουν σχολείο σε σχέση με τα αγόρια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυξάνεται αυτό το ποσοστό και μάλιστα κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά με πολύ βραδείς ρυθμούς. Σύμφωνα με την UNESCO στην υποσαχάρια Αφρική στο γυμνάσιο πηγαίνουν από το κορίτσια το 10% παλιά μέχρι και 35% αυτή τη στιγμή αλλά σε κάθε περίπτωση υπολείπεται πολύ από το 42% των αγοριών οι οποίοι πηγαίνουν τακτικά στο γυμνάσιο, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην υποσαχάρια Αφρική. Δεν θέλω να σας παρουσιάσω όλα τα στοιχεία της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών, αλλά εν ό,τι έχει να κάνει με την απασχόληση, το να πηγαίνουν στο σχολείο, ε, την επιχειρηματικότητα, την υγεία γύρω από το τοκετό και τη γέννηση, την υγεία των μητέρων, είναι τεράστιες οι ανισότητες για όλα αυτά τα θέματα μεταξύ ε, κλινού άστεως και υπαίθρου μεταξύ ε, γυναικών κλπ. Επομένως, ε, θέλουμε να υπογραμμίσουμε τις προτεραιότητες βάσει των ελλημάτων που έχουν διαπιστωθεί και τα πέντε βασικά σημεία που προβάλλω είναι τα, είναι τα εξής. Πρώτον, αφού τα Ηνωμένα Έθνη θα επαναπροσδιορίσουν τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιοετίας, τότε είναι σημαντικό κατά την άποψή μου τουλάχιστον ένας από αυτούς τους στόχους να συνδέεται με τα φύλλα και με τη διάσταση του φύλου. Η ισότητα των φύλων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο σε αυτό το στόχο αλλά και στους υπόλοιπους τέσσερις και σε, μέσα σε κάθε γενικό στόχο να έχουμε επιμέρους στόχους, στόχους καλύτερα εστιασμένους. Τι σημαίνει αυτό. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες είναι τα ε, ε, πρώτα θύματα της υπέρτατης και απόλυτης φτώχειας και τους στερούνται των δικαιωμάτων τους. Επομένως η φτώχυνση, αν θέλετε, των γυναικών έχει δραματικές επιπτώσεις στην διατροφή ε, των ατόμων που εξαρτώνται από τις γυναίκες, παιδιά κολοπού. Και ε, εάν για παράδειγμα πάρουμε τον, ένα γενικότερο στόχο και σε αυτόν έχουμε έναν επιμέρους στόχο των παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο, τότε εάν αυξήσουμε το, ε, του, τους στόχους και ε, έχουμε ποσοτικοποιημένους συγκεκριμένους στόχους για τα κορίτσια, πόσα περισσότερα κορίτσια θα πρέπει να πάνε στο σχολείο, τότε θα μειωθεί ακόμα περισσότερη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών που πηγαίνουν στο σχολείο και αυτό θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο. Από εκεί και πέρα. Δεν έχουμε μόνο ποσοτικούς στόχους, έχουμε και ποιοτικούς στόχους για το 2015 και μετά. Οι δείκτες είναι εξαιρετικά ποσοτικοί ποιοτικού χαρακτήρα, ενώ η φτώχεια είναι μια πολυδιάστατη υπόθεση. Ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δεν έχουν ληφθεί υπόψη μέχρι αυτή τη στιγμή. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, η βία κατά των γυναικών. Ναι, είναι απαραίτητο αυτό. Αλλά όταν υποδεχόμαστε τις γυναίκες που είναι θύματα βίας, στα νοσοκομεία, στα αστυνομικά τμήματα, ο αστυνομικός που παίρνει την κατάθεση έχει καταρτιστεί αυτό είναι ποιοτική διάσταση, δεν είναι ποσοτική. Π.χ. Ε, οικιακή βία μπορεί να κατευθεί το θύμα στις απαραίτητες και ακατάλληλες αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό είναι ποιοτικό στοιχείο επίσης. Ε, πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση γενικότερα. Δηλαδή, οι ποιοτικέ διαστάσεις του θέματος δεν είναι παρούσες σε όλα αυτά τα προγράμματα συνεργασίας και για την ανάπτυξη και το καθεξής. Από εκεί και πέρα, Βασική τομείς και εκεί έχουμε ε, ανάγκη να έχουμε φιλόδοξους στόχους για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των γυναικών σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και πιστεύω ότι η ε, τομείς παρέμβασης είναι αρκετά ευρύς και δίδεται μεγάλη αυτονομία στους αρμοδίους για την εφαρμογή όλων αυτών των προγραμμάτων συνεργασιών πάντοτε με στόχο την ανεξαρτησία και την προσωπική άνθηση των γυναικών, κάτι το οποίο στερούνται πάρα πολλές. Τέταρτον, για να έχουμε όλο και μεγαλύτερη ισότητα των φύλων, οι δωρητές, οι πιστότριες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο, απολύτως απαραίτητο, το λέω και το ξαναλέω, η χρηματοδότηση να συνδέεται με πολύ συγκεκριμένα προγράμματα. Θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση στα προγράμματα που καταπολεμούν την ανισότητα των ε, φύλων. Εγώ είμαι απολύτως πεπισμένη ότι όλοι θα κερδίσουμε αν βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των λαών των αναπτυσσόμενων χωρών πάντοτε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ημών και ημών. Τέλος, μία πρόταση η οποία εξαρτάται από τη συνεργασία μας με την Επιτροπή της ανάπτυξης θα μας επιτρέπει να βάλουμε δεσμευτικές και μη δεσμευτικές ρήτρε για τη μη ύπαρξη διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων στις συμβάσεις που έχουμε τις διμερείς με αυτές τις χώρες. Έτσι θα αναλάβουν αυτές οι χώρες περισσότερες ευθύνες θα εφαρμόσουν περισσότερες κανόνες, θα τίνουν προς την ισότητα των φύλων σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας τους, εάν οι διεθνείς διμερείς τους εμπορικές συμβάσεις περιλαμβάνουν τέτοιου είδου διαστάσεις, τη διάσταση των ισότητας στο φύλων κτλ. Ε, ζητώ συγγνώμη που ε, ε, ε, έφτασα αργά, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι στη διάθεσή σας και με χαρά θα ακούσω τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κανονικά θα μιλούσατε πρώτο και ύστερα θα σας απαντούσαν, όμως όπως είπα το κάναμε αντίστροφο αυτή τη φορά. Συγγνώμη. Υπάρχουν σχόλια σε αυτά που μόλις είπε η συγκήτρια. Έχετε κάτι να πείτε πάνω σε αυτά που μόλις ακούσατε. Όχι από ό,τι φαίνεται. Θα σας πω λοιπόν την προθεσμία για τροπολογίες, τελευταία ημέρα, 25 Φεβρουαρίου. Στις 5 το απόγευμα θα ψηφίσουμε στις 20 Μαρτίου, η Επιτροπή ΔΕΒΕ θα ψηφίσει τον Απρίλιο και θα πάει το θέμα το Μάιο στην Ολομέλεια. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το σημείο αυτό και ολοκληρώνουμε και τη δουλειά μας για σήμερα. Εξαιρετικά νωρίς, πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμενα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αύριο στις 10 το πρωί. Θα σας δω λοιπόν αύριο στις 10. Ευχαριστώ.